evening Καλησπέρα σε όλους. Θα έχουμε μια πολύ σύντομη συνεδρίαση, πολύ ιδιαίτερη. Βλέπω ότι... Ότι είστε εδώ οι περισσότεροι. Έχουμε μόνο τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, για να ψηφίσουμε για τον πρόεδρο της Επιτροπής Είστε σύμφωνοι με την ατζέντα. Όπω είπα, στόχο τη ε, συνεδρία τη αυτή είναι να εκλέξουμε τον πρόεδρο αυτή τη ίδια επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό και προχωράμε λοιπόν άμεσα στην εκλογή. Καταρχά, πρέπει να δούμε τους, ε, ποια μέλη είναι αναπληρωματικά Έχουμε για το Έλκα, έχουμε την Ανιέ Σεβράν και τον Φούλβιο Ματουσέλο που αντικαθιστούν ο τον Ότμαρ Κάρας και ο δεύτερος την Ντανούτα Χούπνερ. S&D, η Βέρα Τάξ αντικαθιστά τον Πολ Τάγκ, στο Ρενιού η Μόνικα Σεμέντο αντικαθιστά τον Ζουλιέ Μποέρ και ο Στεφάν Σεζούρ τον Λουί Πορίτ από τους Πράσινους κανείς από το ECR, ο Μπόγκτα Ρόνσαν, τον ε, κύριο Ντεκούτχο. Ο Νικόλας Αλαβάνος αντικαθιστά τον κύριο Χάμπετ. Και η κυρία Μπίσχοφ, τον κύριο Μαυρίδη από τους σοσιαλιστές. Άλλος ακόμα. Μάλιστα, εγώ αντικαθιστώ τον Πέντρο Σίλβο Φερέιρα, και ονομάζομαι Πέντρο Μάρκες. Μάλιστα το σημειώνουμε. Έχουμε τώρα, παρουσιάσαμε τους ε, ε, αναπληρωτές, τώρα πρέπει να επικυρώσουμε ότι έχουμε απαρτία. Πρέπει να έχουμε 50 μέλη και έχουμε φτάσει αυτή την απαρτία. Λοιπόν, τώρα υποψηφιότητες ε, για την Προεδρία από την πολιτική ομάδα Ποιο θέλει το λόγο, παρακαλώ. Thank you so much. I am glad to communicate. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εξ ονόματο της ομάδα μου να ανακοινώσω την πρόταση τη Σιρένε την άλλη ως νέας Προέδρου της Επιτροπής μας. First of all, Madam. Μάλιστα. Κυρία άλλη δέχεστε την υποψηφιότητα. Να σημειώσω ότι η υποψήφια είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής ΕΚΟΝ και επίσης έχει ολοκληρώσει τη δήλωση συμφερόντων και την δήλωση που έχει να κάνει με την, ε, τον κώδικα διοντολογίας και συμπεριφοράς. Διαβοής μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε ή θέλετε μυστική ψηφοφορία. Όχι. Διαβοής λοιπόν να σας συγχαρώ τότε. So, uh, so madam, please uh, Παρακαλώ λοιπόν να με αντικαταστήσετε εδώ στο Προεδρείο. με χαρά θα εργαστούμε μαζί σας και σας δίνω την θέση σας. Yes. Thank you. Thank you very much. I know that uh, it's a special session. Σας ευχαριστώ. Ε, ξέρω πως ήταν ειδική αυτή εδώ η συνεδρίαση. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο αν έχετε κάτι στα διάφορα και να σας πω πότε είναι η επόμενη μας συνεδρίαση. Καλά, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, εμπιστοσύνη σας και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Έχουμε πολλά, ε, πολλές ενδιαφέρουσες προκλήσεις μπροστά μας και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε αγαστά προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειών που εκπροσωπούμε. Ελπίζω πως θα έχουμε έτσι ένα ευχάριστο κλίμα όπου θα μπορέσουμε να εργαστούμε για το συμφέρον των κρατών μελών μας και των περιφερειών μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να σας ενημερώσω για την επόμενή μας συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα τη Δευτέρα στις 23 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι και την ε, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 9 με 12.30 και 2.30 με 6.30. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ. Πέρα τη συνεδρίαση.